κατέβασε μια τροποποίηση, ένα κείμενο το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάσει του άρθρου 231, συγγνώμη, παράγραφος 4 του κανονισμού, αυτή η τροποποίηση θεωρείται ότι εγκρίνεται, εκτός και αν εντό 24 ερών από την ανακοίνωση, μια πολιτική ομάδα ή αριθμός ευρωβουλευτών, οι οποίοι βασίζονται στο μέσο όρο, δεν θα ζητήσουν ψηφοφορία. Η τροποποίηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας και ο τίτλος θα δημοσιευθεί στα πρακτικά της παρούσας